και που θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ισχυρή βάση, ισχυρά θεμέλια στην Ευρώπη που θα προστατεύουν τους πολίτες. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ κυρία Φερέιρα. Και έτσι λίγη εδώ η κοινή συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το μεσημέρι στις 12.00. Και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, που είναι η προφορική ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Νομισματική Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτική ε, Σταθεροποίηση και η Μελλοντική Δράση. Από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων έχουμε λάβει τον κατάλογο των ε, όσων συμμετέχουν και τα ονόματα αυτών που θα συμμετάσχουν. Η κυρία Sharon Bowles θα λάβει τον λόγο για πέντε λεπτά παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ πολλά τα ζητήματα σήμερα όπου η έκφραση, ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες, αναφέρεται συχνά. Εδώ όμως ο χρόνος ε, δεν μας επιτρέπει να καταλήξουμε σε, σταθερά συμπεράσματα, διότι οι αγορές αποδεικνύουν ότι συνεχώς χρήζουν παρακολούθησης λόγω των εξελίξεων και ότι δεν μπορούμε να έχουμε διαρκή και μόνιμα συμπεράσματα. Είναι πολλές οι δοκιμασίες που αποδεικνύουν ότι χρειάζομαστε διαφανείς προτάσεις αλλά και αποτελέσματα που να δημοσιεύονται. Έτσι λοιπόν καθυστερήσαμε πολύ για να φτάσουμε στην λεπτομέρεια του σχεδίου διάσωσης της Ελλάδας. Και η Επιτροπή καθυστερούσε για μήνε μέχρι να επεξεργαστεί τι λεπτομέρειε. Εμεί είμαστε λοιπόν οι διάβολοι που κοιτάζουμε τι λεπτομέρειε και καθυστερούμε. Στι 11 Μαου ο Μηχανισμό Ευρωπαϊκή Σταθεροποίηση προβλέφθηκε και άρχισε να λειτουργεί χρησιμοποιώντα τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό ω πηγή του. Χρειάστηκε τόσο πολύ καιρό για να καταλήξουμε σε υποσχέσει που είχαμε αναλάβει νωρίτερα που αυτό δεν έφτανε. Έτσι στι 7 Ιουνίου το γενικότερο, η γενικότερη διευκόλυνση χρηματοπιστωτική ε, δημιουργήθηκε και άρχισε να λειτουργεί. Εδώ θα αν είχαμε βιαστεί λίγο περισσότερο θα ήμασταν ίσως πιο αποτελεσματικοί και πιο φτηνοί. Τώρα, για τα αποτελέσματα της λειτουργίας από των δύο εργαλείων, των μέσων για τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και για την δανειοδότηση άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, όπως της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων. Εδώ θα έχουμε σίγουρα καλά αποτελέσματα ε, και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το κρατικό χρέο ευρωπαϊκών κρατών, δανείζοντα τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Γιατί η πραγματική οικονομία είναι αυτή που πληρώνει το τίμημα των οικονομικών κρίσεων. Τι θα γίνει λοιπόν με το μετριασμό τέτοιων φαινομένων, γιατί η ανάπτυξη είναι τόσο σημαντική για την ανάκαμψη και οι μικρομεσαίε επιχειρήσει θα μα βγάλουν από τη σημερινή κρίση. Ο σκοπό των μέσων αυτών είναι να ενισχύσει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Διότι χώρε που δεν βρίσκονται στην Ευρωζώνη και θέλουν να προσχωρήσουν στον μηχανισμό αυτό θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν. Οι κανόνε ε, του μηχανισμού έχουν αλλάξει προκειμένου να είναι ευνοϊκέ ω προ αυτό. Πραγματικά, γενικότερα, όπω αποφασίστηκε και χθε στην Επιτροπή, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την παρακολούθηση των ισολογισμών και τα κάτι μελη να φροντίσουν για το θέμα αυτό, προβλέποντα τα απαραίτητα μέτρα. Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα που παραμένουν εκρεμή. Πώ θα καθοριστεί ο συντονισμό μεταξύ του Ταμείου Σταθεροποίηση και του πώ λειτουργεί το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο εάν θα προβληθούν κονδύλια διετήλογου χάρη ανάλογα με τις αιτήσει που υποβάλλονται και ποια θα είναι η σχέση μεταξύ των επιτοκίων ε, στη μια και στην άλλη πλευρά τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Νομισματικού Ταμείου θα δίνονται με τους ίδιους όρους ή θα είναι αποκλειστικά τα δάνεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε περίπτωση αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων των ε, δανειοληπτών θα πρέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις διάσωσης ή αυτό να το κάνει ο μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει ο μηχανισμός να δραστηριοποιείται αμέσως ή πρώτα απ' όλα να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Να κοιτάξουμε τώρα τα ευρωομόλογα. Υπήρξε ένα σημαντικό ζήτημα που έπρεπε να μας απασχολήσει εδώ και αυτό ήταν το γενικότερο ζήτημα των ευρωομολόγων σε σχέση με τα σημερινά επικοινωνία τόκια. Διότι για τη φορολογική πειθαρχία, για τι αγορέ. ήταν ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα αυτό ώστε να το σέβονται οι δυνάμει τη αγορά. Όμω αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα φαίνεται ότι θα είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα του χρέου πολύ νωρίτερα αν είχαμε αναλάβει δράση για τα, κρατικά, για τα ομόλογα αυτά. Το κρατικό χρέο, οι κεφαλαϊκέ απαιτήσει και η σχετική οδηγία έπρεπε να έχουν ήδη λειτουργήσει τα επικίνδυνα ομόλογα και οι, δυνα... οι αποκλήσεις δανειστικές είναι κάτι που έπρεπε να έχει ληφθεί υπόψη. Δεν θα πρέπει πάλι να διασώσουμε τις τράπεζες μέσω του μηχανισμού σταθεροποίησης όπως είχε γίνει πρόσφατα. Γιατί ε, οι δοκιμασίες πίεσης που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον θα πρέπει να είναι λιγότερο πιεστικές. Η κοινή οικονομική διακυβέρνηση μας δείχνει ότι πρέπει να προβλέψουμε επισκευές συνολικές για το μέλλον. Και να έχουμε μια διαδικασία αντιμετώπισης του ελλείμματος που όμως δεν μας επιτρέπει να υπολογίσουμε και σε μηδενικούς κινδύνους. Εδώ έχουμε την ευκαιρία ένα πρόβλημα από την ε, οδηγία κεφαλαιοκικών απαιτήσεων να το μετατρέψουμε σε εργαλείο χρήσιμο για το μέλλον. Έτσι λοιπόν εκφράζω την ικανοποίησή μου που η Επιτροπή υπέδειξε την πρόθεσή της να ε, συμμετέχει με το Κοινοβούλιο σε συζητήσει για την οικονομική διακυβέρνηση και την εποπτεία στι ερχόμενε νομοθετικέ τη προτάσει. Η Επιτροπή μα αναπομονεί να συμμετάσχει ενεργά σε αυτή την ε, συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ, Σάρων Μπόου. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει τον λόγο. Ο Επίτροπο Μπάρνιε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα αντιληφθήκατε ότι επειδή αποουσιάζει ο συνάδελφο Ρεν, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσω περισσότερο χρόνο στην τελική μου απάντηση. Αναφέρθηκε η κυρία Μπόλου σε αγγέλους. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άγγελοι όταν μιλάμε για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες από την κυρία Μπόλουσου ότι όντω ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες και θα φροντίσω να απαντήσω όσο πιο λεπτομεριακά γίνεται. Πρώτα απ' όλα περί ποιου ποσού πρόκειται όταν μιλάμε για αυτό τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίησης και ποιο είναι η σχέση με το ανώτατο όριο των ίδιων πόρων. Τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Κοφέιν αναφέρθηκαν σε 60 δις ευρώ για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το και το 2.2 του κανονισμού 407 αναφέρει ότι τα δάνεια περιέχονται στο ανώτατο όριο των ίδιων πόρων και εδώ περιορίζονται τα ποσά σύμφωνα με απόφαση των μελών και ανέρχονται σε 1,23% του ε, ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή το συνδυασμένο το συνδυασμό ανώτατο όριο είναι το σύνολο των κονδυλίων που, προσφέρονται, που θα προσφέρουν για την εξυπηρέτηση του χρέου δεν πρέπει να ξεπερνάνε το 1,23% κατά τη διάρκεια ενός ε, οικονομικού έτους. Αυτή είναι μια δήλωση του Όλη Ρέντε. Διάβασα. Ε, τώρα η Κομισιόν θα κάνει μια εκτίμηση αντικτύπου τώρα, σύμφωνα με τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίησης η Κομισιόν είναι υποχρεωμένη εντός εξαμήνου μετά από τη σύσταση αυτού του μηχανισμού ε, και κάθε έξι μήνες μια έκθεση λειτουργία. Αυτό το κείμενο θα υπολυθεί στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και θα αναφέρεται στην λειτουργία αυτού του ευρωπαϊκού ε, μηχανισμού χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Τρίτο ερώτημα. Τι επιπτώσεις θα έχει στις δημοσιονομικές ικανότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Δεν θα έχει καμία άμεση επίπτωση στις δραστηριότητες ε, χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ε, η ρευστότητα θα παραμείνει ως ε, έχει ανεπηρέαστη από τον μηχανισμό αυτό. Δεν ε, θα δανείζει εξ ονόματος ε, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η ΕΤΕ. Τώρα, ένας παρόμοιος μηχανισμός και με και σε ποια νομική βάση θα λειτουργήσει. Η Κομισιόν εργάζεται σε στενή συνεργασία με την ομάδα εργασία τη οποία ε, προεδρεύει ο πρόεδρο Βαν Ρομπέη. Η διαδικασία τη επιλογή μάλλον τη νομική βάση δεν έχει γίνει. Οπότε, ποιο θα είναι ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται για κάθε εξέλιξη σε ό,τι φορά το σύνολο αυτών των νέων διαδικασιών. Η νομική μορφή συμμετοχή του Κοινοβουλίου θα εξαρθεί από την νομική βάση που θα έχουμε όπως σύμφωνα με τι ε, συνθήκες. Τώρα, με ποιο τρόπο θα λειτουργήσει ο συντονισμό μεταξύ Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση ε, κλπ. Θα λειτουργήσει λοιπόν σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πακέτο, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού αλλά και του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Έβδομη ερώτηση. Πώ θα ανταποκριθείτε σε μια ανάγκη χωρών που δεν είναι μέλη του ευρώ, ε, τα κράτη-μέλη τα οποία δεν ε, ε, συμμετέχουν στον μηχανισμό της Ευρωζώνης ε, θα μπορούν να κάνουν αναφορά στην, στην, προσφυγή τους, ε, του άρθρου για την χρηματοπιστωτική στήριξη. Ήδη έχουν δεσμευτεί 15 δις για δάνεια προς τη Ρουμανία, τη Λετωνία και την Ουγγαρία. Εξάλλου, συνθήκες δανειοδότησης αφορούν στο ισοζύγιο πληρωμών και με τρόπο ιδιαίτερα ευνοϊκό από ό,τι προβλέπεται στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τώρα και τέλος, το άρθρο 122.2 της συνθήκης χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τον κανονισμό, για αυτόν τον μηχανισμό σταθεροποίησης διότι το Συμβούλιο και η Κομισιόν ενήργησαν ε, σε κάτω από συνθήκες επίγουσες διότι οι χώρες απειλούνται από σοβαρές εξελίξεις που οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα που εξέβηγαν του ελέγχου τους. Η Κομισιόν λοιπόν ενήργησε άμεσα προκειμένου να προστατεύσει το ευρώ. Θα ήταν δύσκολο λοιπόν να συμβαστεί με μια χρονοβόρα διαδικασία η οποία θα, στην οποία συμμετείχαν και κάποια εθνικά κοινοβούλια. Ε, τον προσθέτω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει από την Κομισιόν σε ένα ψήφισμα τον Απρίλιο 2009 να υιοθετήσει κανονισμό για τη βοήθεια προ τα κράτη-μέλη με βάση ακριβώ αυτό το άρθρο 122 τη συνθήκη. Αυτά έχω να σα απαντήσω, κυρία Μπόλ, σχετικά με τα συγκεκριμένα ερωτήματα που είχατε θέσει. Ευχαριστούμε θερμά κύριε Επίτροπε. Και τώρα περνάμε στους αγορητέ εξ ονόματο των κοινοβουλευτικών ομάδων. Ο κύριος Ορμακάρας πρώτος για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. 1,5 λεπτό κύριε Κάρας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Πρώτον, δυστυχώ τώρα δεν μπορώ την περιφρόνηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου και του κανονισμού να είμαι ιδιαίτερα ευγενής. Όμως θα ήθελα να επικεντρωθώ στο θέμα ο μηχανισμός σταθεροποίησης αντικαθιστά πιστεύουμε την δημιουργία δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου και Εποπτείας. Χρειαζόμαστε τα πρώτα βήματα για την δημιουργία του ιδίου κεφαλαίου για μια ευρωπαϊκή ε, έναν ευρωπαϊκό οίκο αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Η σταθεροποίηση και οι μηχανισμοί σταθεροποίησης ε, των αγορών δείχνουν πόσο κατεπίγουσες είναι οι ανάγκες μεταρρύθμισης ε, των αγορών. Δείχνει επίσης και την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός μηχανισμού για την κρίση. Δείχνει όμως ότι σε σχέση με την οικονομική Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε και μια πολιτική ένωση και μια πιο αποτελεσματική οικονομική ένωση. Η καλύτερη σταθεροποιητική μηχανή είναι η τήρηση των κριτηρίων του Μαστρίχτ, η τήρηση των κριτηρίων της, ε, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, μέσα στην πραγματικότητα της ε, αγοράς και μια πολιτική για τον ανταγωνισμό που θα βασίζεται σε μια επιθετική δράση και δραστηριοποίηση και για να διασφαλίζεται η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να μην παίρνουμε χρήματα από τους φορολογούμενους που θα πληρώνουν τα σπασμένα. Ευχαριστώ θερμά για την ε, συμμαχία ε, των Δημοκρατών. Η κυρία Ποδηματά θα λάβει τον λόγο παρακαλώ. Δύο λεπτά. Πολύ, κυρία πρόεδρε κύριε επίτροπε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η απόφαση τη 9 η μαου για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοπιστωτική σταθεροποίηση ήταν καθοριστική σημασία για την προστασία του ενιαίου νομίσματο και γενικότερα τη σταθερότητα τη ζώνη του ευρώ. γι' αυτό και το κοινοβούλιο το οποίο είχε ζητήσει προπολού από το συμβούλιο να προχωρήσει προ αυτή την κατεύθυνση τη χαιρέτησε άμεσα η απόφαση αυτή όπως και η απόφαση για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διευκόλυνσης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας έστειλαν τελικά έστω και καθυστερημένα ένα μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης της ευρωζώνης προς τις διεθνείς αγορές. την ίδια ετοιμότητα και αλληλεγγύη έδειξε και η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα με την απόφασή της για προσωρινή παρέμβαση στη δευτερογενή αγορά ομολόγων πρακτική η οποία συνάδει πλήρως με το γενικότερο πνεύμα της απόφασης των υπουργών οικονομία της ζώνης του ευρώ. πρόκειται ωστόσο για μηχανισμούς και μέτρα προσωρινού χαρακτήρα και αν θέλουμε πραγματικά να αντλήσουμε διδάγματα από τη σημερινή κρίση είναι προφανές ότι δεν πρέπει να περιμένουμε την επόμενη κρίση να αναδείξει ξανά τις ελλείψεις και τις αδυναμίες της ευρωζώνης και της ένωσης για να αποφασίσουμε να παρέμβουμε. σήμερα είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσουμε στη δημιουργία μόνιμων μηχανισμών οικονομικού συντονισμού και εποπτείας που θα λειτουργούν όχι μόνο κατασταλτικά αλλά κυρίω προληπτικά στο πλαίσιο αυτό η πρόσφατη ανακοίνωση τη Επιτροπή για την ενίσχυση του οικονομικού συντονισμού είναι ασφαλώ προ τη σωστή κατεύθυνση. δεν θα πρέπει όμω να ξεχνάμε ότι ο βασικό μα στόχο είναι η σταθερή και βιώσιμη ανάκαμψη τη Ευρωπαϊκή οικονομίας και γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο οικονομική διακυβέρνηση που δεν θα εστιάζει μόνο στον πυλώνα τη δημοσιονομική εξυγίανση αλλά και στην προστασία τη απασχόληση, στην ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή. για να το πετύχουμε προτεραιότητά μα δεν πρέπει να είναι κυρώσεις αλλά τα κίνητρα και τα μέτρα πρόληψης που θα διασφαλίζουν την ισότιμη μεταχείριση όλων των κρατών μελών της ένωσης και των πολιτών τους. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα η άλλοι εγγεγραμμένοι ομιλητές. Η κυρία Μπερές, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, γνωρίζετε ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρόμαστε ε, που πριτάνευση η αλληλεγγύη, παρόλο που είναι κρίμα που χρειάστηκε να περάσουν ε, τόσοι μήνες μετά την πρωτοβουλία του Προέδρου Χέρμαν Ρομπό για τη σύγκληση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 11 Φεβρουαρίου για το θέμα αυτό και στο μεταξύ οι αγορές έκαναν τη δουλειά τους. Κατά την εξέταση αυτής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης θα πρέπει να κοιτάξουμε και το παρελθόν, να δούμε από πώς δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση επειδή δεν είχαμε αρκετά στοιχεία χρηστής διακυβέρνησης στη ζώνη ευρώ. Ο Ότμαρ μίλησε για το Σύμφωνο Σταθερότητας. Έχω την αίσθηση ότι η εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας δεν αρκεί. Και φαίνεται ότι υποτιμήσαμε από την αρχή τους κινδύνους απόκλησης σε ό,τι αφορά τα δημόσια χρέη. Σήμερα έχουμε έναν μηχανισμό που θεσπίστηκε σε μια έκτακτη περίπτωση και λίγο Τώρα, από τον Οκτώβριο του 2008, από την εφαρμογή του μηχανισμού, ζητήθηκε το άρθρο 122 να αναλυθεί περαιτέρω. Έγινε κάπως εκτάκτος ε, και βιαστικά φυσικά η βιασύνη δεν είναι ο καλύτερος σύμβουλος πάντα. Βέβαια, είπαμε ότι ίσως υπάρχει καλύτερη λύση από τη διαιώνιση αυτού του μηχανισμού. Ελπίζω να καταθέσετε πιο επιθετικές προτάσεις στον τομέα αυτό, γιατί είμαστε βέβαιοι ότι μια ζώνη σαν τη ζώνη ευρώ χρειάζεται όχι μόνο μια χρηστή διακυβέρνηση για να αποσοβηθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον, αλλά σε περίπτωση που ανακύψουν και πάλι στο μέλλον χρειαζόμαστε έναν ε, ισόβιο, ένα μόνιμο μηχανισμό. Επίσης, τα κράτη-μέλη, αντί να ε, προτιμούν το μηχανισμό το Special Purpose Vehicle ή τα ευρωμόλογα, να δουν πώς ε, λειτουργούν τέτοιου είδους δομές στην αγορά. Και απατώντας την κυρία Σαρομπόλ, ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δυστυχώς ε, η πρόεδρος διακόπτη την κυρία Μπέρες. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Δύο λεπτά χρόνο είχατε, δυόμιση μιλήσατε. Ωραία. Καλή διαδικασία, να κάνουμε έτσι καλύτερα, για να έχουμε χρόνο και να τηρούμε και τους κανόνες και κανείς να μην χάνει το χρόνο ομιλία του. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Πάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Μπαζέσκου, για ένα λεπτό έχει πρώτη το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Στις 9 Μαΐου, οι Υπουργοί Οικονομικών των κρατών μελών αποφάσισαν τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού ε, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που εντάσσεται σε ένα πακέτο μέτρων που στόχο έχουν την προστασία του ενιαίου νομίσματος, του ευρώ και την ε, ανόρθωση της οικονομικής κατάστασης των κρατών μελών. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να χρησιμοποιείται με αποτελεσματικό τρόπο σε περίπτωση που τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να εξηγιάνουν με δικές τους προσπάθειες τα οικονομικά τους. Και από την άποψη αυτή ε, βοηθούν τα κράτη-μέλη για να επανέλθουν σε μια, υγειονομική, ε, μια υγιή, υγιή χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Βέβαια, διανύσαμε μια κρίση για την οποία δεν ήμασταν προετοιμασμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Μπαρνία, δεδομένου του προσωρινού χαρακτήρα του μηχανισμού αυτού, που είναι τριετή και δεδομένη τη ανάγκη που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδρά ταχύτατα και άμεσα σε περιπτώσει ε, κρίσεων, δεν πιστεύετε ότι είναι καλύτερη η λύση η διαιώνιση αυτού του μηχανισμού και ποιο πιστεύετε ότι είναι ο κατάλληλο μηχανισμό για κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή, ο κύριο Όμπερμαϊερ, για ένα λεπτό πάλι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σε περίπτωση κρίσης κράτους μέλους, τα άλλα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να βοηθούν με άμεσα δημοσιονομικά πακέτα, αλλά να κρύβονται. Ακούγεται καλά ή να εγγυώνται, συγγνώμη. Ε, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα αυτό, γιατί η Ευρωζώνη αρχίζει να παρουσιάζει μεγάλες ανισότητες και αυτό είναι μεγάλη, μεγάλο πρόβλημα, το οποίο και αυτο ειναι μεγαλο προβλημα το οποιο αναβαλλεται Ο δε πολίτης γρήγορα γίνεται ο φιλέτης. Επίσης ε, είναι το θέμα της εξάρτησης από οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Θα πρέπει λοιπόν να ε, λαμβάνεται υπόψη το, η αξιολόγηση από αυτές τις ε, ε εταιρείες που είναι ε, αμερικανικής βάσης ως επιτοπλίστων. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν και ε, άλλες δυνατότητες και όχι μόνο ε, οι ιδιωτικές αυτές ε, εταιρείες αξιολόγησης. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε να μην συσσωρεύονται τα χρέη όλων μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Ρούμπικ έχει το λόγο τώρα για ένα λεπτό πάλι. Κυρία Πρόεδρε Κοχμέριν και Επίτροπε Μπαρνιέ, για μένα τίθεται το θέμα της σταθεροποίησης και της οικονομικής μεγέθυνσης. Το ερώτημα είναι ότι ο προϋπολογισμός για το 2011 είναι διαπραγμάτευση. Ξέρετε γραμμές του προϋπολογισμού που θα ενισχύσουν την απασχόληση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πώς μπορούν να υποστηριχθούν με καλύτερο τρόπο και πώς θα έχουμε καλύτερους ε, περισσότερους επιχειρηματίες. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της σταθεροποίησης. Γιατί όταν ε, αυξηθεί η οικονομία θα μπορούμε να έχουμε καλύτερη διανομή και δικαιοσύνη. Το πρόγραμμα ε, ΣΥΠ για τον ανταγωνισμό και την ε, καινοτομία θα μας ε, βοηθήσει πάρα πολύ. Μια περικοπή, όπως προβλέπετε τώρα για το πρόγραμμα αυτό, είναι εντελώ αντιπαραγωγική πιστεύω. Στην ανάλυση μας πρέπει να προσέξουμε ποιες γραμμές του προϋπολογισμού ε, υποσκάπτουν την απασχόληση, ποιε είναι ουδέτερε και ποιε δημιουργούν καλύτερη απασχόληση. Θα περιμένουμε πρόταση από εσά. Και τώρα η κυρία Μπερές πάλι για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά ε, την τράπεζα, ε, το θέμα είναι να δούμε σε ποια περίπτωση και υπό ποιου όρους θα μπορεί να προχωρεί σε δανειοδοτήσεις ε, στην αγορά και με βάση και τους ε, συντελεστές. Και θέλω να θέσω ένα ερώτημα στον Επίτροπο. Στο πλαίσιο αυτό ε, τι πιστεύετε στο πλαίσιο της ομάδα εργασίας υπό τον Χέρμαν von Ρομπάι, μήπως θα έπρεπε να γίνει πρόταση ή ο Επίτροπος Ρεν ενδεχομένως, θα έπρεπε να διατυπώσει πρόταση να εξεταστεί η αμοιβεοποίηση ορισμένων ε, από τα κυρίαρχα αυτά χρέη. Είναι ένα θέμα βέβαια εκτός πεδίου αρμοδιοτήτων αυτής της ομάδας εργασίας, αλλά νομίζω ότι στο πλαίσιο των προτάσεων που υπάρχει πέτος να διποθούν, αυτή η πρότασή μου νομίζω ότι θα έπρεπε να διατυπωσει προταση να εξεταστει η αμοιβεοποιηση ορισμενων απο τα κυριαρχα αυτα χρεη ειναι ενα θεμα βεβαια εκτος πεδιου ορμοδιοτητων αυτης της ομαδα εργασιας υπόψη wieder die Kommission das Wort. Herr Kommissar Barnier, bitte schön. Euh, si vous euh, σε ό,τι αφορά το πολύ σημαντικό ζήτημα για τα ευρωομόλογα και τα τελευταία σημεία τα οποία ανέφερε η κυρία θα σας απαντήσει φαντάζομαι απευθείας ε, εντός των προσεχών ημερών εγγράφος ο αρμόδιος επίτροπος ο κύριος Ρένης. Ό,τι αφορά την ε, αρχική παρέμβαση για τις δοκιμές αντοχής αν θέλετε ή κοπόσεως σε περίπτωση ε, που προκύψουν, ίσως δεν προκύψουν βέβαια αντίστοιχα φαινόμενα, θα πρέπει να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νωρί και ο πρόεδρος Μπαρόζα εξέφρασε και τη δική του άποψη, όπως και όλοι Ρεν, είπαμε ότι η διαφάνεια πραγματικά είναι μεγάλη αρετή και έχει πολλά πλεονεκτήματα. Σας παραπέμπω λοιπόν στα σχόλια του Προέδρου της Επιτροπής κ. Μπαρόζο. Ο κ. Κάρα τώρα ανέφερε ένα σημείο ιδιαίτερα σημαντικό που το είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη συζήτηση για την πρόληψη και συγκεκριμένα ότι οι τράπεζες είναι αυτές που πρέπει να πληρώνουν για τις τράπεζες και όχι φορολογούμενοι. Επιβεβαιώνω ότι στην ανακοίνωσή μου θα δώσουμε βάρος στο θέμα αυτό. Ε, θα έχουμε τη σχετική νομοθεσία από το 2011 και θα υπάρχει ο σχετικός μηχανισμός πρόληψης ή ε, επίλυση ώστε πρόληψη η αντίστοιχη αρχή ο ρηπαίνων πληρώνει. Και γνωρίζουμε ότι κάλιον το προλαμβάνει παρά το θεραπεύουν. Κοστίζει λιγότερο η πρόληψη. Σε ό,τι αφορά αυτή την εισφορά, την τραπεζική εισφορά, είναι ένα εργαλείο. Ενδέχεται να υπάρξουν και άλλα. Ο ρηπαινων πληρωνει και γνωριζουμε οτι κάλλιον το προλαμβανει παρα το θεραπευουν κοστιζει λιγοτερο η προληψη σε οτι αφορα είναι να μπορούμε να ταυτοποιούμε τους κινδύνους έγκαιρα πριν μεταβληθούν σε κρίσεις που θα μεταβληθούν με τη σειρά σε καταστροφές. Θα εξετάζουμε λοιπόν ε, όλα τα ζητήματα, είπε και η κυρία Μπερές μεταξύ άλλων ε, για τα κυρίαρχα χρέη και τη βαθμολόγησή τους. Θέλω να σας πω ότι πράγματι θα επεξεργαστούμε και το ζήτημα αυτό, τη διαφοροποίηση αγορών που κάποιες φορές είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένες αν θέλετε και θα δούμε και για το, το ενδεχόμενο την επιλογή ενός ευρωπαϊκού οργανισμού. Όλα αυτά θα μεταφραστούν σε μια νομοθετική πρόταση τέλη 2010, αρχές 2011. Η κυρία Μπερές πάντα, η οποία ανέφερε την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας, συμφωνώ και εγώ μαζί σας, πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη πιο μακριά. Είπατε και το έχετε καταλάβει καλά ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο μηχανισμός χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης, παντός συγχρόνως και στην κυρία Μπαζέσκου. Ε, θέλουμε πράγματι έναν διαρκέστερο, έναν πιο ισόβιο ε, μηχανισμό. Σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας υπό τον κύριο Φαντρομπάη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει βέβαια ακόμη επιλέξει την νομική βάση, αλλά θα διατυπώσουμε σχετικές προτάσεις ε, για έναν πιο μόνιμο μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ε, για την κυρία Ποδηματά το έργο το οποίο επιτελείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το γνωρίζετε πολύ καλά. Η Ελλάδα έχει αναλάβει μια σημαντική δέσμευση. Ε, η ελληνική κυβέρνηση πρέπει και αυτή να βάλει το δικό της λιθαράκι στην προσπάθεια αυτή. Σίγουρα η χώρα σας ε, επλήγει από αυτή την κρίση πάρα πολύ σοβαρά μάλιστα. Σίγουρα δεν θέλουμε να θέσουμε που στην ανεξαρτησία των κρατών μελών, ιδίω των κρατών μελών τη Ευρωζώνη. Πάντω ε, έγινε ακόμη πιο αναγκαίο ε, το να δείχνει κανεί αποφασιστικότητα για να παίρνει τα διορθωτικά μέτρα ώστε να μην πληγεί η Ευρωζώνη στο σύνολό τη. Και το ΕΚΟΦΗΝ ε, στις 9 Μαΐου ε, που αποφάσισε τη δημιουργία αυτών των δύο μηχανισμών νομίζω ότι απέδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δράσει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις μεγάλες αυτές οικονομικές προκλήσεις. Σίγουρα χρειάζεται μεγαλύτερος συντονισμός ε, οικονομικός και χρηματοπιστωτικός μπορεί κάποιο να θεωρεί παροχημένο τον όρο συντονισμό, πρέπει να περβούμε ακόμη και το συντονισμό και να κάνουμε ακόμη ένα βήμα ε, προ τα εμπρό. Πάντω, ε, νομίζω ότι έχουμε ήδη αντλήσει διδάγματα και δεν έχουμε ε, φτάσει ακόμη στην έξοδο του τούνελ. Θα αντλήσουμε και άλλα διδάγματα από όλες αυτές τις αναταράξεις και για το ευρώ και για την Ελλάδα με προτάσεις διακυβέρνησης, με προτάσεις συντονισμού για ένα σύστημα λοιπόν ε, ανταπόκρισης, αντίδρασης και σταθεροποίησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει και σημαντικές προτάσεις ό,τι αφορά την δημοσιονομική επιτήρηση και εποπτεία Ούτε αυτά όμως αρκούν. Πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερα πράγματα γιατί οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, περιμένουν από εμάς να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις για την ανάπτυξη και για την απασχόληση. Μιλάμε λοιπόν για διακυβέρνηση, μιλάμε για σταθεροποίηση, μιλάμε για προσπάθειες, για ρύθμιση. Νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και για ανάληψη πρωτοβουλίας στο επίπεδο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για να επανέλθουμε στην ε, αύξηση της απασχόλησης ε, και της ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου μου λοιπόν, ε, μαζί με 10 συναδέλφους μου, θα σας ε, υποβάλω σχετική πρόταση αρχές Οκτωβρίου για το λεγόμενο Single Market Act, την πράξη της ενίας αγοράς. Έτσι θα έχουμε λοιπόν την πλατφόρμα, αν θέλετε, τη βάση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η ενιαία αγορά των 500 εκατομμύριων πολιτών με πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θέλουμε να διαψεύσουμε τις ελπίδες όλων αυτών των πολιτών. Θα πρέπει η ενιαία αγορά να υπηρετεί τον πολίτη να υπηρετεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θέλουμε να αυξήσουμε τα ποσοστά ανάπτυξης. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα λέμε και πρέπει να τα μεταφράζουμε και σε συγκεκριμένες πράξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ υπευλήθη από την Επιτροπή την Οικονομική και Νομισματική την Νομισματική Επιτροπή ένα κείμενο ε, Β70318